Colleghi. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ε, ξεκινήσουμε τις ε, εργασίες μας, γιατί με τον τρόπο αυτό θα τιμήσουμε και τους συνάδελφου εκείνους οι οποίοι ήρθαν στην ώρα τους. Το πρώτο λοιπόν σημείο είναι η έγκριση της ε, ημερήσιας ε, διάταξης. Ε, φαντάζομαι θα έχετε λάβει υπόψη σας τις τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα χθε το πρωί. Αυτές κοινοποιήθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Αυτές λοιπόν οι αλλαγές αφορούν το ότι στις 11 θα προτάξουμε το θέμα για την Αλγερία σήμερα. Μετά το τέλος συνειδήσης θα έχουμε ψηφοφορία και επίσης αύριο το πρωί θα ψηφίσουμε για την έκθεση Λίζεκ. Υπάρχει λοιπόν μια νέα ημερήσια διάταξη η οποία υπάρχει μόνο στα αγγλικά. Αυτή η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει αυτές τις αλλαγές τις οποίες ε, και σας ανέφερα. Φαντάζομαι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Πολύ ωραία. Προχωράμε. Δεύτερο σημείο αφορά την έγκριση των πρακτικών ε, τη συνεδρία 22 Σεπτεμβρίου, τη 4η Οκτωβρίου, τη 11η Οκτωβρίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, ε, α ε, θεωρήσουμε ότι τα πρακτικά αυτά εγκρίνονται. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Τρίτο σημείο. Σχέδιο έκθεσης ε, που περιέχει πρόταση σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προ το Συμβούλιο σχετικά με μια συνεκτική πολιτική έναντι των αυταρχικών καθεστώτων κατά των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα όταν αυτά προωθούν τα προσωπικά και εμπορικά του συμφέροντα εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πρόκειται για την δεύτερη εξέταση σύστασης πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εφαρμοστεί μια ε, συνεπής πολιτική απέναντι σε αυτά τα αρχικά, ε, αυταρχικά καθεστώτα έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει περιοριστικά μέτρα. Ο εισηγητής είναι ο Σερ Γκράχαμ Βότσον. Στις 5 Οκτωβρίου κατέθεσε την πρόταση σύστασης ε, και ένας εμπειρογνώμονας έκανε επίσης μια σύντομη μελέτη των κυρώσεων που μπορούν να ληφθούν απέναντι σε μια σειρά χωρών. Θα ήθελα λοιπόν να σα υπενθυμίσω ότι στις 17 Οκτωβρίου εξέπνευσε η προθεσμία για την κατάθεση ε, των τροπολογιών και κατετέθησαν 139 τροπολογίες. Θα ήθελα λοιπόν ο κύριος Βότσεν να σχολιάσει αυτές τις τροπολογίες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους σας. Ελπίζω ότι δεν θα χρειάζεται να καταδαπανίσω πολύ από το χρόνο σας σήμερα. Όπως είπε και ο Ερίκος ο Όγδος σε μία από τις έξι γυναίκα του, γυναίκες του, την Άνε, την Άν Μπολέν, της είπε «Δεν μην στενοχωριέσαι, δεν θα σε κρατήσω για πάρα πολύ». Λοιπόν, είναι μια μεγάλη χαρά να παρουσιάσω για δεύτερη φορά Ε, νομίζω ότι αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα εργασία. Ο James Madison στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάλι ποτέ ο μεγάλος φεδεραλιστής, ίσως θα χαιρόταν πολύ για όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε για να οικοδομήσουμε μια κοινότητα αξιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτό το πνεύμα σας φέρνω αυτή την πρόταση για ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής σε σχέση με τις κυρώσεις, που θα πρέπει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι καθεστώτων τα οποία ως αυταρχικά είναι αντικείμενο περιοριστικών μέτρων. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι στο φως της συζήτησης που είχαμε και μετά την εξέλιξη αυτή της συζήτησης θα ήταν χρήσιμο να αλλάξουμε και την επικεφαλίδα της έκθεσης και να λέει ο τίτλος αυτός πρόταση για μια σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σε σχέση με μια συνεκτική πολιτική έναντι καθεστώτων για τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα όταν οι ηγέτες τους ασκούν τα εμπορικά και άλλα οικονομικά τους συμφέροντα εκτός, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή να μην υπάρχει μνήμα αυταρχικών καθεστώτων και να αναφέρεται ότι πρόκειται για καθιστότητα έναν των οποίων ήδη εφαρμόζουμε κάποιο είδους περιοριστικά μέτρα. Και φυσικά, κύριε Πρόεδρε, οι συνάδελφοι δεν χρειάζεται να τους υπενθυμίσω ότι μετά από τα γεγονότα <clears throat> της Αραβικής Άνοιξης φέτος, όταν βρεθήκαμε ουσιαστικά έκθετη λόγω της υποστήριξής μας για κάποιους από τους δικτάτορες της Βόρειας Αφρικής που τώρα έχουν εξοβελιστεί από τους αγανακτισμένους πολίτες τους, η έκθεση αυτή είναι και επίκαιρη για το λόγο αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους συναδέλφους για την προσοχή που έχουν δώσει στην έκθεση αυτή και για τις τροπολογίες που έχουν υποβάλει. Επίσης να ευχαριστήσω τη γραμματεία, ιδίως τον Μάρκο Αλόνσο για την υποστήριξή του και τη βοήθεια που μου έδωσε για να μπορέσω να ομαδοποιήσω αυτές τις τροπολογίες και να τις αντιμετωπίσω με τροπολογίες συμβιβασμού και επίσης και τους κύριους εισηγητές για το θαυμάσιο έργο το οποίο φέρασε σε πέρας για να με αρρωγήσουν στο να μπορέσω να επιτύχω μια ευρεία <clears throat> συνένεση για την έκθεση αυτή. Ίσως χρειάζεται να κάνω και δύο διευκρινήσεις. Καταρχήν, σε σχέση με τη χρήση του όρου κυρώσεις από τη μία πλευρά και περιοριστικά μέτρα, περιοριστικών μέτρων από την άλλη πλευρά. Στις συνθήκες της η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναφέρεται πουθενά σε κυρώσεις. Μιλάμε για περιοριστικά μέτρα. Οι κυρώσεις είναι ένας όρος των Ηνωμένων Εθνών. Όταν εφαρμόσουμε αυτές τις, ε, κυρώσει μέσω των Ηνωμένων Εθνών, τις ονομάζουμε περιοριστικά μέτρα, αλλά πολλές φορές εφαρμόσουμε δικά μας περιοριστικά μέτρα, τα οποία δεν έχουν εγκριθεί σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Αυτός είναι ο λόγος και για τον οποίο θα ήθελα να προτείνω να μην δεχτούμε την τροπολογία 43 που ζητά ένα σαφή ορισμό. Δυστυχώς, στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο όρος κυρώσεις δεν εμφανίζεται πουθενά. Η δεύτερη διευκρίνηση που θέλω να κάνω αφορά το ρόλο που ζητούμε να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε στη φάση οικοδόμησης της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας που θα πρέπει να υπηρετήσει αυτή η υπηρεσία. Εγώ πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει και κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής περιοριστικών μέτρων και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση αυτών των μέτρων. Δεν είναι ο στόχος μου το Κοινοβούλιο να παίζει ρόλο σε οποιαδήποτε λήψη απόφασης σε σχέση με το ποια περιοριστικά μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν εναντίον ποιου και πότε. Αυτό πιστεύω ότι είναι το έργο των διοικητικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε τις περισσότερες τροπολογίες, τη μεγάλη πλειοψηφία των τροπολογιών, σε 16 συμβιβαστικές τροπολογίες. Ο κίνδυνος είναι πάντα σε μια τέτοια διαδικασία ότι καταλήγουμε σε μια σύσταση η οποία είναι σαν μια κουρελού ή σαν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν συνάφεια κατά ανάγκη με τα υπόλοιπα. Ο στόχος μας όμως θα πρέπει να είναι να κρατήσουμε σαφή το στόχο αυτού του, αυτής της σύστασης και ελπίζω οι συνάδελφοι να το έχουν υπόψη τους όταν φτάσουμε στην έγκριση του εγγράφου αυτού και την ψήφιση των τροπολογιών ότι πρέπει να διατηρήσουμε τη συνεκτικότητά του. Πολύ ωραία. Πριν λοιπόν δώσω το λόγο στους ε, σκιώδεις εισηγητές ε, και σε όλους τους αδέλφους που επιθυμούν να λάβουν το λόγο, θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω να τοποθετηθείτε στην πρόταση που έκανε ο εισηγητής σχετικά με την κατάργηση τις ε, λέξεις αυταρχικών καθεστώτων του επιθέτου πριν από τα καθεστώτα. Αυτό περιλαμβάνεται στην επικεφαλίδα της έκθεσης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, εγκρίνουμε την πρόταση του εισηγητή κυρίου Βότσον. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Από ό,τι βλέπω όχι. Πολύ ωραία. Τώρα, σκιώδεις εισηγητές, συνάδελφος Τζάγκλ και ελπίζω Γέγκλε, η κυρία Γέγκλε, η Γερμανίδα, αλλά δυστυχώ, λέει ο πρόεδρο ε, δεν πρόφερα σωστά το όνομά της. Παρακαλώ, κυρία Γέγκλε. Πολύ σωστά, κύριε Πρόεδρε, και σα ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή μας ε, για την έκθεσή του, για την ε, ειλικρίνεια ε, για τον ε, τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε τις ε, τροπολογίες και τις συμπεριέλαβε σε συμβαστικές προτάσεις. Εγώ, εκ μέρους των συναδέλφων του ΕΛΚ. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω ε, γιατί πραγματικά υπήρχε πνεύμα συνεργασίας και όπως το είπε και ο εισηγητής Πράγματι, ο στόχος είναι να υπάρχει ε, διευκρίνηση του σκοπού, να μην έχουμε ένα κατάλογο, μία λίστα επιθυμιών για τα Χριστούγεννα. Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε. Θα το καταφέρουμε αν συνεχίσουμε τον δρόμο που έχουμε χαράξει. Για μας λοιπόν, για το ΕΛΚ, είναι σημαντικό σε όλες τις ε, δραστηριότητες ε, τις οποίες αναπτύσσουμε απέναντι σε τέτοια καθεστώτα να έχουμε πάντα κατά νου μας τους πολίτες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εξάλλου, ε, θα μου επιτρέψει να πω και το εξής. Πρέπει λιγάκι να ξανασκεφτούμε τις λέξεις που έχουμε επιλέξει, ε, κυρώσεις, τις λέξεις κυρώσεις και τις λέξεις περιοριστικά μέτρα. Αυτό ήδη το είπαμε και χθες. Ε, επειδή γνωρίζουμε ποιοι είναι οι ορισμοί, ε, παρόλα αυτά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται σε προγενέστερο στάδιο. Δηλαδή όχι το σύνολο των περιοριστικών μέτρων, να μην αποφασίζουμε για αυτό το σύνολο, αλλά σε μια προγενέστερη φάση να συζητάμε ενδεχομένω για την επιβολή κυρώσεων και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το διευκρινίσουμε μεταξύ μας. Κατά τα άλλα, ε, για μας είναι σημαντικό, συμπεριλαμβάνεται εξάλλου στην έκθεση, το ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου και πάντα την φάση που ακολουθεί, το μετά, δηλαδή το πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε εμείς σε θέματα οικοδόμησης κράτους δικαίου, εκδημοκρατισμού μιας χώρας, ε, παροχή βοήθειας ε, σε εκλογές. Αυτός είναι ο στόχος και η βούληση της ΕΛΚ. Δηλαδή δεν πρέπει να ε, σπάμε τελείως τις σχέσεις με τις χώρες αυτές, να τις διαταράσουμε παντελώς, να αφήνουμε πάντα ένα παράθυρο ανοιχτό για σε τελική ανάλυση και η οικονομική συνεργασία είναι κάτι που μας ε, ενδιαφέρει. Αυτό το οποίο επίσης είναι σημαντικό είναι το εξής. Επειδή υπάρχουν στρατηγικά, οικονομικά συμφέροντα, επειδή υπάρχουν και ιδεολογικά συμφέροντα, δεν θα πρέπει να εφαρμόζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Νομίζω ότι όσον αφορά το θέμα αυτό, συμφωνούμε όλοι μας. Για άλλη μια φορά λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω ότι για το θέμα αυτό θα καταλήξουμε σε μια σαφή σύσταση, έτσι ώστε και εμείς ως Κοινοβούλιο να διεκδικούμε το σεβασμό που μας προσήκει. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ε, το λόγο τώρα θα ήθελα να δώσω στο συνάδελφο Τσάλα από τους ε, σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος διότι και μπορώ να εκτιμήσω τις συμβιβαστικές τροπολογίες, θα τις εξετάσουμε εξετάζονται σε αυτή την έκθεση είχα δύο βασικά μελήματα σχετικά με την, την έκθεση. Πρώτον, για την εκπαίδευση για τα παιδιά των ξένων ηγετών. Νομίζω ότι το λύσαμε αυτό το πρόβλημα πολύ απλά. Αποφύγαμε αυτή τη διατύπωση και τονίσαμε ε, πολύ περισσότερο το θέμα της απαγόρευσης, της ε, θεώρησης, ε, και με, αυτό το σύστημα μπορέσαμε να καλύψουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι προσπαθούμε να ποσοτικοποιήσουμε κριτήρια ε, για τα μέτρα και το καθεστώς κυρώσεων, πότε πυροδοτείται το καθεστώς κυρώσεων. Νομίζω ότι αποφύγαμε αυτήν τη διατύπωση και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και στις άλλες τροπολογίες μπορέσαμε να επιτύχουμε κάποια ισορροπία ανάμεσα στις ευθύνες του Κοινοβουλίου και τις ευθύνες της εκτελεστικής εξουσίας και νομίζω ότι για μια τέτοιου είδους έκθεση αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι καμιά φορά αναμειγνύονται οι αρμοδιότητες μας και οι ευθύνες μας. Νομίζω είμαι έτοιμος να υποστηρίξω όλες τις συμβιβαστικές τροπολογίες, όπως και τις περισσότερες από τις άλλες τροπολογίες που κατέθεσε ο εισήγητης και οι συνάδελφοι από τις άλλες πολιτικές ομάδες, διότι νομίζω ότι ενισχύουν σημαντικά την εισήγηση αυτή και το πνεύμα αυτής της εισήγησης. Ευχαριστώ πολύ. Grazie. La parola al signor James Συνάδελφος James Key Bright από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ίσως άρχισαν και ορισμένα σχόλια. Θα ήθελα να πω εν συντομία ότι όπως ανέφερα την τελευταία φορά, απαντώντας σε μια πρόσκληση από την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας. Προσπαθούμε να αναθεωρήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και ως μέρος αυτού αναφέρθηκε η παρακολούθηση πολύ συχνά από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι σημαντικά και αυτό νομίζω έχει σχέση με τη συζήτησή σας. Θέλω επίσης να προσθέσω ότι όπως είπε και η κυρία Γέγλε, οι κυρώσεις αποτελούν μέρος ενός πακέτου μέτρων και πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη το πολιτικό περιεχόμενο και τα άλλα μέτρα που ισχύουν. Ε, ε, ήμουν ικανοποιημένο από αυτήν τη συζήτηση τελευταία φορά και είναι ενδιαφέρον το ότι η συζήτησή σας απηχεί μερικές από τις ε, παρατηρήσεις που εκφράσαμε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ασφάλειας για την αναθεώρηση των βελτίστων πρακτικών. Κοιτάξτε, σα ζήτησα να παρέμβετε εσεί να λάβετε το λόγο, γιατί ε, δεν είχαν ζητήσει άλλοι συνάδελφοι το λόγο και γι' αυτό το λόγο σα έδωσα ήδη τώρα, αν θέλετε, το λόγο. Τώρα, ο εισηγητή ε, επιθυμεί να απαντήσει, παρακαλώ. Ε, δεν έχω πάρα πολλά πράγματα να προσθέσω. Θα ήθελα απλά να ξαναευχαριστήσω ε, την κυρία Γίγκλε και τον κύριο Τσάλα για την αρρωγή τους, ε, όπως επίσης και τους άλλους ε, σκιώδης που και αυτοί διευκόλυναν τη δουλειά μου, με διευκόλυναν στο να επιτύχω τη συνένεση σε ένα θέμα τόσο σημαντικό. Τώρα. Στα αγγλικά. Για να απαντήσω αυτά που είπε ο κύριος <clears throat> Κιμπράιτ, Εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά τα οποία ανέφερα. Νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα τομέα ο οποίος θα απαιτήσει περαιτέρω συζητήσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και των αρμοδίων αρχών της εκτελεστικής εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο διαμορφώνεται η, εξωτερική, η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας αλλά ελπίζω ότι θα είναι σαφής ο στόχος μας και η εκτελεστική εξουσία δεν θα λησμονήσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δείξει μεγάλη, ε, μεγάλο ενδιαφέρον και μέρημνα στο να υπάρχει συνεκτικός χαρακτήρας στην επιβολή αυτών των κυρώσεων βάσει μιας κλιμάκωσης προτεραιοτήτων και μέτρων που μπορεί να εφαρμοστεί σε κυβερνήσεις οποιασδήποτε χώρας ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη σημασία τους, ή την πολιτική κατεύθυνση των ηγετών τους, ώστε να είναι σαφές ότι δρούμε επί τη βάση αρχών και όχι ότι ουσιαστικά όταν έχουμε να κάνουμε με ισχυρές και μεγάλες χώρες ότι κάπου αφήνουμε κατά μέρο τις ανησυχίες μας. Αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι σαν μια δύναμη για δημοκρατία στον κόσμο θα πρέπει να είναι φανερό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι φαίνεται να εφαρμόζει μια πολιτική που να βασίζεται σε σαφείς αρχές και ελπίζω ότι αυτό θα προκύψει <clears throat> ως αποτέλεσμα και της αίτησης της πολιτικής και Επιτροπής Ασφάλειας για να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Πολύ, ωραία. Σας ε, υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία για αυτή την πρόταση ψηφίσματος θα είναι ε, στις 20 Δεκεμβρίου στην επόμενη συνεδρίασή μας. Ε, και πραγματικά ε, σας συγχαίρω για τα τελικά σας κύριε Βότσον. Πάρα πολύ ωραία τα τελικά σας. Προτείνω λοιπόν να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να περιμένουμε τον επόμενο ο τον κύριο Κόβατσεφ. Πολύ ωραία συνάδελφοι, μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και πάλι τις εργασίες μας ε, στο επόμενο θέμα που αφορά στην τροποποίηση του κανονισμού 539 κάθετος 2001 του Συμβουλίου ε, που αναφέρει τον κατάλογο των τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινε στην υποχρέωση θεώρηση ε, για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου των τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε ε, στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και επ' αυτού θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Κόβατσεφ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, χαιρετίζω την πρόταση της Κομισιόν για την ε, τροποποίηση του κανονισμού 539 2001. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τον κατάλογο των τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρηση για τη έλευση των εξωτερικών ιστορών των κρατών μελών και τον κατάλογο των τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Είναι ο θετικός και ο αρνητικός κατάλογος. Όπως αναφέρεται και τον, ε, στην αρχή πρέπει να υπάρξει επικαιροποίηση της αμοιβαιότητας έτσι ώστε να υπάρχει ε, και ε, εφαρμογή της ιδρυτικής συνθήκης της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει σημαντικότερο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη ρήτρα διασφάλισης η οποία αυτή τη στιγμή προβλέπει την εξαίρεση κάποιων χωρών. Νομίζω ότι η, Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μια ευελιξία εφόσον κριθεί απαραίτητο για κάποιες χώρες για τις οποίες υπάρχουν επιφυλάξεις ε, κυρίως σε θέματα μετανάστευσης. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα πολύ σημαντικό που αφορά τη στάση Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε άλλες χώρες. Όσον αφορά την ύπαρξη αυτή τη ρήτρα διασφάλισης αυτή η ρήτρα προσφέρει ένα πλαίσιο για το μέλλον και αυτό το πλαίσιο μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να ξεπεραστεί η διστακτικότητα ορισμένων κρατών μελών, να ανοίξει ο δρόμος για την άρση θεωρήσεων και με τον τρόπο αυτό να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στο μηχανισμό λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως για θέματα τρίτων χωρών. Θα ήθελα λοιπόν να στηρίξω αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα κράτη-μέλη ε, να παρουσιάσουν ε, κάποια επιχειρήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν πρέπει να υπάρχει αυτοματισμός. Δεν μπορεί αυτόματα να αναστέλλεται ε, προσωρινά το σύστημα μη υποχρέωση θεώρησης για ορισμένες χώρες πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγησης ε, που θα έχει σχέση με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτές τις τρίτες χώρες, αλλά και γενικότερα απέναντι στην περιοχή στην οποία βρίσκονται αυτές οι τρίτες χώρες. Σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να περιλάβουμε ε, και τις πληροφορίες που παίρνουμε από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Τη σχετική τροπολογία έχω ε, συμπεριλάβει στην πρότασή μου. Όσον αφορά τώρα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, εγώ έχω να προτείνω μία ε, τροπολογία που ε, την επισήμανα και στους αδέλφους στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Οι προτάσεις των συναδέλφων, οι περισσότερες από αυτές πρέπει να στηθούν στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και δεν θα αποφασιστούν από εμάς. Εγώ λοιπόν περιμένω να ακούσω την άποψη και τα σχόλια των συναδέλφων. Τάνια Φαγιόν, η συνάδελφος ε, η οποία είναι σκιώδη συγγήτρια των ε, σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω σλοβένικα. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το σχέδιο αυτό το οποίο παρουσίασε ο εισηγητής μας. Πρέπει να πω ότι εδώ πρέπει να αποφασίσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο από πολιτική έποψη. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι μονάχα ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά ξέρουμε όλοι ότι το θέμα της ελευθερίας διακίνησης είναι υποαπειλή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι υπήρξε και πίεση κατά της ζώνης του Σέγγεν και της συμπερίληψης χωρών στην περιοχή αυτή. Η πρόταση αυτή δημιουργήθηκε μετά από το πρώτο κύμα προσφύγων από την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων που προσπαθήσαν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο παράνομο. Επομένως είναι ένα ευαίσθητο πολιτικά θέματα. Εγώ έχω επομένως από τη μία πλευρά θετική αντιμετώπιση για την ε, θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προσωρινά μέτρα για τη μη χορήγηση βίζας, αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να υπόκειται σε μία ανάλυση, σε μία ενδελεχή ανάλυση για να πραγματοποιηθεί. Εγώ φοβάμαι στην πραγματικότητα θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, ότι ορισμένε χώρε θα χρησιμοποιήσουν αυτή την κατάσταση για να εξυπηρετήσουν πολιτικούς σκοπούς. Θέλω λοιπόν να εκφράσω εδώ τι ανησυχίε μου. Βάσει της πρόταση Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει μονάχα ένα συμβουλευτικό ρόλο. Εδώ δεν ακολουθείται η διαδικασία η οποία ίσχυε στο παρελθόν για ένα τέτοιο κανονισμό. Η Κομισιόν στο παρελθόν δεν ήταν υποχρεωμένη ούτε το Συμβούλιο να λαμβάνει υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου. Εγώ πιστεύω ότι η Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τύχουν κοινή πληροφόρηση για οποιοδήποτε θέμα που ανακύπτει και να έχουν μία εβδομάδα για να σταθμίσουν τη θέση τους. Επίσης, σε σχέση με τα ποσοστά τα οποία αναφέρονται, βάσει της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί οποιοδήποτε κράτος μέλος να εφαρμόσει ένα σύστημα με το οποίο αναστέλλεται το σύστημα παροχής προξενικών θεωρήσεων και εφαρμόζεται ένα κατόφλι 50% στη συνέχεια. Στην αρχή φαίνεται ότι αυτό το 50% είναι πολύ υψηλό, αλλά ήδη στην προηγούμενη δεκαετία η Γερμανία έχει εφαρμόσει μέτρα αυτού του είδους. Εδώ δίνεται υπερβολική ελευθερία στην ε, Κομισιόν και στα κράτη-μέλη για την άρση του καθεστώτος αυτού. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της αιτιολόγησης μιας τέτοιας απόφασης. Εδώ δεν πρέπει να μιλάμε για ποσοστά, αλλά για σημαντικές μέσα στο χρόνο αυξήσεις του αριθμού των ετούντων ασύλου που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση ε, μεταναστών ή προσφύγων σε μία ή σε κάποια άλλη χώρα αλλά πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο στη διαδικασία αυτή και η Επιτροπή Δημοσιολευθεριών συγκεκριμένα. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να υπάρξει και συμφωνία των δύο επιτροπών στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο και δεν μπορεί να παραγωνίζεται σε σχέση με την προσωρινή εφαρμογή μιας άρσης του καθεστώτος ε, προξενικών θεωρήσεων. Τίθενται λοιπόν πολιτικά ερωτήματα για τη ρήτρα διασφάλισης και εγώ πιστεύω ότι να λάβετε υπόψη και τις προφορικές τροποποιήσεις που έχω διατυπώσει χθε. Ελπίζω ότι όλα αυτά θα βοηθήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τονίσει ότι πρέπει να υπάρχει ένα καθεστώς εξαίρεσης από την υποχρέωση προξενικής θεώρησης απαλλαγής για τις χώρες αυτές των Δυτικών Βαλκανίων που έχουν κάνει σημαντικά βήματα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα απαραίτητα τεχνικά κριτήρια, αλλά θα πρέπει να δώσουμε και το κατάλληλο μήνυμα προς τις χώρες αυτές ότι είμαστε σοβαροί σε σχέση με τη θέση μας. Argentini, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, στα πρόσφατα έτη, ή μάλλον θα το εκφράσω διαφορετικά, τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε την Αραβική Άνοιξη και σε αυτό το Κοινοβούλιο είχαμε συζήτηση σχετικά με τους τινήσιους που καταφεύγουν στην Ευρώπη και φοβούμε ότι η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί και θα παραταθεί. και θα λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις και θα πυροδοτήσει φόβους σχετικά με τις θεωρήσεις σε άτομα που έρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέμε ότι θέλουμε την απελευθέρωση του συστήματος των θεωρήσεων, αλλά είναι κάτι το οποίο φοβούμε. Συμφωνώ με την ε, κυρία Φαγιόν. Θα πρέπει να σκεφτούμε πιο προσεκτικά, με περισσότερη σύνεση, γιατί ίσως θα πρέπει να είμαστε λιγότερο φιλελεύθεροι σχετικά με τις ε, θεωρήσεις και να λάβουμε υπόψη τις ε, μεταναστευτικές ροές και να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και πώς, και ε, η πολιτική των θεωρήσεων έχει επιπτώσει στην εξωτερική μας ε, πολιτική, στους γείτονές μας. Νομίζω ότι αυτή η τροπολογία είναι καλή τροπολογία και ελπίζω ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα κάνει μια τέτοια ε, πρόταση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ πολύ. Bene, altri interventi? Πολύ ωραία. Επιθυμεί κάποιο άλλο παρακαλώ να λάβει το λόγο. Από ό,τι φαίνεται όχι. Κατόπιν τούτου θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον βέβαια επιθυμεί να παρέμβει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοβατσέφ για το σχέδιο εισήγησής του που νομίζω είναι πολύ καλή εισήγηση, την χαιρετίζουμε με ενδιαφέρον σχετικά με την τροπολογία που προτάθηκε από τον κύριο Κοβατσέφ. Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε ότι έχει νόημα και ε, είναι σημαντικό να περιλάβουμε αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε τέτοιες αποφάσεις. Αν θα πρέπει να ξαναεπιβάλλουμε δηλαδή την υποχρέωση θεώρησης όσον αφορά και την επανεισδοχή. Ωστόσο, υπάρχει κάτι ε, που είναι θεσμικό. Δεν ξέρω πώς η υπηρεσία εξωτερικής δράσης το αντιμετωπίζει και το Κοινοβούλιο σε αυτές ε, τις ε, τροπολογίες από θεσμικής απόψεως, αλλά νομίζω ότι πρέπει το θέμα αυτό να διευκρινιστεί, αλλά η ιδέα είναι δεκτή από εμά. Σχετικά με την τροπολογία της κυρίας Φαγιόμ, θα ήθελα να πω ότι το θέμα το οποίο έθεσε εκεί είναι σημαντικό, σχετίζεται με τον ρόλο του Κοινοβουλίου. Εμείς στην δική μας πρόταση έχουμε προτείνει αυστηρά κριτήρια ότως ώστε ε, να πυροδοτείται η ρήτρα διασφάλισης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νομίζω την επιτροπολογία η οποία είναι απαραίτητη και νομίζω ότι σε τέτοιες σε περιπτώσεις ε, κατεπίγουσας ανάγκης ε, θα πρέπει να μπορούμε να λάβουμε γρήγορα τέτοιες αποφάσεις. Μιλούμε για την επιτροπολογία. Πρέπει να δίνουμε στο Κοινοβούλιο μία εβδομάδα για να δίνει την συνένεσή του την έγκριση του προτού υιοθετήσουμε ή εφαρμόσουμε μια απόφαση. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι σύμφωνο προς την Επιτροπολογία και μπορεί να θέσει ένα πρόβλημα από θεσμικής απόψεως. Νομίζω λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε το θέμα αυτό με προσοχή ακόμη και μόνο από τη θεσμική πλευρά. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω με την ευκαιρία αυτή ότι η Επιτροπή δεσμεύθηκε να παρέχει πλήρεις πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για ενδεχόμενη πυροδότηση ε, του, της ε, ρήτρας διασφάλισης, αυτό λέγεται στην αιτιολογική έκθεση, δεν έχουμε καμία πρόθεση να αφήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτός μιας τέτοιας απόφασης. Αν, να, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την επιτροπολογία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για αυτά που κάνουμε από θεσμικής απόψεως. Όσον αφορά τα ποσοστά, όπως έχουμε ήδη πει, ε, την 66 βεβαίως νομίζω ότι εσείς θέλετε να το συζητήσουμε. Αυτό το θέμα έχει συζητηθεί και στο Συμβούλιο με τα κράτη-μέλη, η Επιτροπή και πάλι. Αν ε, μπορούμε να έχουμε την επιτροπολογία και δεν χρειαζόμαστε ποσοστά, η Επιτροπή θα μπορούσε να δεχτεί αυτή την κατάσταση, αλλά το βασικό για μας είναι η επιτροπολογία την οποία χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι θα αρκεστώ σε αυτά τα σχόλια για την ώρα. Βεβαίως, και πάλι θα ξανασυζητήσουμε το θέμα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ πολύ. Εισηγητά, θέλετε κύριε Σιγητά να λάβετε το λόγο, να απαντήσετε. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την, την ε, Κομισιόν και τον κύριο εισηγητή στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ όπου συζητήσαμε για τη διαδικασία αυτή, <clears throat> την εισηγητρία συγκεκριμένα. Εγώ συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας αλλά νομίζω ότι αναπόκειται στην Επιτροπή Δημοσίου Ελευθεριών να αποφασίσει για τα ποσοστά, για τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα κράτος μέλος ή περισσότερα για να κοινοποιήσει μια έκτακτη κατάσταση μετανάστευση στην Κομισιόν. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα Δυτικά Βαλκάνια. Ξέρουμε πολύ καλά όμως γιατί έχει διατυπωθεί αυτή η πρόταση. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λοιπόν, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία επιτροπολογίας, για τη λήψη απόφασης. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για το αν θα εξασφαλιστεί και η συμμετοχή του Κοινοβουλίου μέσα σε ένα χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας ώστε να γνωμοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγκεκριμένα η Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών, φαντάζομαι η Επιτροπή Λίμπε να δώσει γνωμοδότηση για τα θέματα αυτά και η Κομισιόν θα πρέπει να δώσει στο Κοινοβούλιο όλες τις πληροφορίες και όλα αυτά αφορούν μονάχα το ενδεχόμενο μιας προσωρινής αναστολής. Δεν πρόκειται για μια μόνιμη ρύθμιση σε μια χώρα, για μια χώρα η οποία περνάει από τον θετικό κατάλογο στον αρνητικό κατάλογο ή τούμπαλιν. Δεν έχουμε λοιπόν μια τέτοια πρόνοια στο... στην πρόταση αυτή να υπάρξει μια μεταφορά μια χώρα από ένα κατάλογο σε έναν άλλο για το διηνεκές, μόνο σε προσωρινό επίπεδο. Επομένω, ω Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα πρέπει να αποδεχτούμε αυτή την πρόταση και εγώ από την δική μου πλευρά υποστηρίζω αυτά που είπε η κυρία Βέμπα. Όλες οι άλλες προτάσεις όμως θα πρέπει να εξεταστούν από την Επιτροπή ε, Δημοσίων Ελευθεριών, όπως και αυτές. Πολύ ωραία. Σήμερα στις 6 και 4, σας υπενθυμίζω, θα ψηφίσουμε ε, για αυτό το θέμα, για την τροποποίηση του κανονισμού. Επόμενο θέμα, η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα των χωρών BRICS και άλλων αναδειωμένων δυνάμεων, στόχοι και στρατηγικές. Ε, συγκητής, ο κύριος Σάιρους Βόλσκι και ε, θα ήθελα ε, να σας πω ότι για να υπάρχει αρκετός χρόνος για να υπάρξει γνωμοδότηση, η έγκριση της γνωμοδότησης ορίστηκε για τις 20 Νοεμβρίου. Ε, λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τη συνάντηση με τον νέο επικεφαλής αντιπροσωπείας για την Ινδία, που θα λάβει η χώρα στις 11 ε, και 4 ε, για να προλάβουμε όλα αυτά θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σάιρους Βόλσκι να κάνει μια εισαγωγή και σας παρακαλώ πάρα πολύ την εισήγησή να την περιορίσετε σε 5 λεπτά. Uh, Προσπαθήσω να είμαι σύντομος κύριε Πρόεδρο. 10 λεπτά έχετε. Μπορείτε να διπλασιάσετε τον χρόνο σα. Δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει ο κύριο Σάριο Βόλσκι. Θέλω να ευχαριστήσω όλου αυτού που συνέβαλαν με τροπολογίε στην έκθεση αυτή. Είναι πάρα πολύ χρήσιμε αυτέ οι τροπολογίε. Συγχρόνω, οι περισσότερε τροπολογίες υποστηρίζουν τη δική μου θέση, κάτι το οποίο δείχνει και τη σημασία του αντικειμένου που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω όσο το δυνατόν περισσότερο το περιεχόμενο αυτών των 164 τροπολογιών. Είχαμε μια πρώτη συνάντηση σκιωδών ηγητών. και νομίζω ότι συμφωνούν και οι συνάδελφοι ότι είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πλήρη συνένεση για το κείμενο αυτό. Υπήρξε κάποια διαμάχη ίσως στην πρώτη αυτή συζήτησή μας, η οποία μπορεί να ξεπεραστεί Δηλαδή να πούμε ότι από τη μια πλευρά οι χώρες BRICS αξίζουν ιδιαίτερη αντιμετώπισης και προσοχής από την ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά παράλληλα θα πρέπει να κατανοήσουμε την πολυπικιλία των χωρών αυτών. <clears throat> αλλά συγχρόνως αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί με μια προσέγγιση ομαδοποιημένη. Γι' αυτό ζητώ να έχουμε αυτή τη διτή προσέγγιση προς τις χώρες αυτές και από κοινού και μεμονωμένα όταν αυτό είναι απαραίτητο με την κατάλληλη διαδικασία συντονισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν λαμβάνονται κοινέ δράσεις και γι' αυτό απαιτούνται και τα, καλύτερα, τα κατάλληλα εργαλεία εξωτερικής πολιτικής ώστε να προκαταλαμβάνουμε τις, ε, τις ενέργειές τους και όχι απλώς να αντιδρούμε εκ των υστέρων και μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικοδομητική η συμμετοχή τους σε πολλές ενέργειες εξωτερικές πολιτικές Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουν λάβει θέσεις οι οποίες δεν είναι πάντα συμβατές με τις δικές μας θέσεις, αλλά στο Ηνωμένο, στα Ηνωμένα Έθνη πολλές φορές είναι σημαντικό αυτό όταν εμείς θέλουμε να έχουμε μια ενιαία στάση. Δεύτερον για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τρίτον για την κλιματική αλλαγή. Για όλους αυτούς τους λόγους θέλω να υπογραμμίσω ότι χρειάζεται συνεργασία και χρειάζεται να είμαστε να δρούμε ε, εγκαίρως και όχι, να είμαστε προορατικοί και όχι να στρουθοκαμιλίζομεν. Και με το να χώρουμε το κεφάλι μας στην άμμο όσοι στρουθοκάμιλος δεν θα εξαφανιστούν αυτές οι χώρες. Ο στόχος μας δεν πρέπει να είναι να διατηρήσουμε στο κλουβί τους τις χώρες αυτές, αλλά να έχουμε μια έγκαιρη αντιμετώπιση και να κατανοήσουμε ότι μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο οι χώρε αυτέ σε θέματα εξωτερική πολιτική. Αν τι πάρουμε για δεδομένε, αν τι παραγνωρίσουμε, αν δεν αναγνωρίσουμε την ύπαρξή του, θα χάσουμε μια πραγματική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε χρήσιμους εταίρους για τη διαμόρφωση της παγκόσμιας τάξης που είναι και κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και είναι ο κομβικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει λοιπόν να χάσουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε μαζί με τις χώρες αυτές τη νέα παγκόσμια τάξη και να βασιστούμε μαζί τους σε κοινέ δράσεις τη στιγμή που αναδύεται ένα νέο στερέωμα διεθνών δυνάμεων και γι' αυτό θα πρέπει να προετοιμάσουμε στρατηγικές. Αυτό σημαίνει πρέπει να έχουμε και τα κατάλληλα εργαλεία. Δεν ζητώ να υπάρξει μια νέα μονάδα ή ένα νέο τμήμα στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης, αλλά θα πρέπει η ΕΑΔ να λάβει υπόψη της την ανάγκη προετοιμασίας και συντονισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν εν ολίγης οι θέσεις μου και θέλω και πάλι να πω ότι είμαι αισιόδοξο ότι όλες οι τόσο αξιόλογες συνεισφορές των συναδέλφων θα μπορέσουν να ενσωματωθούν στο τελικό έγγραφο της έκθεσης αυτής και προσβλέπω στη συζήτηση με τους σκιώδεις εισηγητές που θα γίνει στις 13 Δεκεμβρίου για να ψηφίσουμε στις 20 Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Ο Τζάλα ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι ήταν ενδιαφέρουσα και ουσιώδη η συζήτηση για τα θέματα αυτά και σε ακαδημαϊκό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο για την προσέγγιση μας προς τις χώρες BRIC. Η έννοια αυτή των χωρών BRIC είναι και το αντικείμενο της συζήτησής μας, μερικές φορές μιλάμε για τις χώρες αυτές σαν να είναι μια ενότητα, σαν ένα ενιαίο σύνολο. Άλλες φορές αντιμετωπίζουμε σαν μεμονωμένες χώρες, πέντε μεμονωμένες χώρες και έχουμε διαφορετική προσέγγιση έναντι αυτών. Αυτό είναι σωστό γιατί πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή στάση για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν πολύ περισσότερες διαφορές παρά ομοιότητες μεταξύ των χωρών αυτών. Και γι' αυτό η συζήτηση μεταξύ μας και σας στόχο να εξεύρει μια ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών προσεγγίσεων, τι ομαδοποιημένες και τις μεμονωμένες, η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία. Ναι, Νότια Αφρική λέω, ο και η Ρωσία. Είναι χώρες που έχουν μεγάλη σημασία. Θα πρέπει να βρούμε κάποια ισορροπία μεταξύ τη στάση μα εναντί των χωρών αυτών. Είναι βέβαια δύσκολο να έχουμε μία ενιαία στάση μαζί τους στα Ηνωμένα Έθνη, γιατί είναι πολλές φορές όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν πάντα μία ενιαία στάση, αλλά το να βρούμε μία ισορροπία είναι πάρα πολύ σημαντικό και το να μην θέτουμε το κεφάλι μας στην άμμο όπως η, η είναι πολύ σημαντικό γιατί οι χώρες αυτές οι BRICS μπορούν να είναι πολύ προβληματικές στα Ηνωμένα Έθνη σε ορισμένα σημεία. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση τους πια για τα, την κλιματική αλλαγή που είναι ένα ανοιχτό θέμα, αλλά πιστεύω και αυτή είναι η δεύτερη μου παρατήρηση, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε νέα εργαλεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι, αυτά θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε μια διμερή στρατηγική εταιρική σχέση. Ίσως μπορούμε να τονίσουμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια διμερή στρατηγική εταιρική σχέση. Είναι σημαντικό αυτό. Και αυτό δεν είναι μονάχα θέμα που αφορά τις χώρες αυτές, τις χώρες BRICS. Όταν μιλάω λοιπόν Χαίρομαι ιδιαίτερα επίσης που μπορώ να υποστηρίξω ορισμένες από τις τροπολογίες των σκιωδών εισηγητών γιατί ενισχύουν την έκθεσή μας και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να εξεύρουμε μια λογική ισορροπία. Έχουμε ένα μήνα περίπου στη διάθεσή μας και είμαι απόλυτα αισιόδοξο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πολυθετικό. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ζάλα, Ο κύριος Σάλα ήταν στη συνεδρίαση ε, και φιλοσόφησε και σκέφτηκα ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνεδρίαση αυτή όταν μιλήσαμε όχι μόνο για τις χώρες BRICS αλλά και για την ποια θα έπρεπε να είναι η στάση της Ευρώπης απέναντι στις χώρες αυτές. Αυτό που φοβούμε και το επαναλαμβάνω είναι ότι ότι πρέπει Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η κατάσταση στον κόσμο αλλάζει. Πρόκειται για αναδυόμενες χώρες οι οποίες αποκτούν όλο και περισσότερη ισχύ εμπνεόμενες από την ιστορία τους, μπορεί να είναι ιστορία απεικιοκρατίας, αλλά πάντως θα έπρεπε να έχουμε μια στάση απέναντι στις χώρες αυτές που να αναγνωρίζει μια καινούρια ισορροπία στον κόσμο και ελπίζω ότι το αποτέλεσμα της φιλοσοφικής μας συζήτησης θα είναι μια έκθεση που θα εκφράζει την ανησυχία των Ευρωπαίων ε, και σχετικά με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να αντιδρά, να απαντά σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται. Γι' αυτό η έκθεση αυτή αφήνει περιθώριο για να προσπαθήσουμε να βρούμε μια καινούρια ισορροπία και να βρούμε τη θέση μας μέσα σε αυτήν την καινούρια κατάσταση, τη νέα ισορροπία. Υπάρχει μεγάλη πρόκληση να ασχοληθούμε με αυτές ε, τις πολυπληθείς ε, τροπολογίες. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε συμβιβασμούς, αλλά αυτοί οι συμβιβασμοί θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη νέα ισορροπία στον κόσμο. Χαίρομαι που μπορώ να συνεισφέρω σε αυτή την εργασία. Συνάδελφος ε, για την Μάκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης είναι ιδιαίτερα ευρύ. Ο συνάδελφος κύριος Σάριος Βόλσκι έχει ενώπιόν του μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική έκθεση. Καταλαβαίνω ότι και ο ίδιος θα ήθελε να εξασφαλίσει τον καλύτερο δυνατό συντονισμό μεταξύ μας γιατί η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυτό το σημαντικό στοιχείο που είναι ακριβώς η σχέση με τις χώρες BRICS. Πρέπει να πω όμως ότι έχω μία κάπως διαφορετική άποψη από τον κύριο Σάριους Βόλσκι. προτού μπω σε αυτό το σημείο όμως θέλω να υπογραμμίσω αυτό το οποίο είπε ο εισηγητής ότι η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι πιο σαφώς τα χέρια της υπάτης εκπροσώπου. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι ουτοπία να μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο ο Υπουργός Εξωτερικών της, των ΗΠΑ και να πάρει στο τηλέφωνο τον υπεύθυνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, η Άγγελα Μέρκελ, η καγκελάριος της Γερμανίας, δεν έχει βοηθήσει πολύ στο να υπάρχει ενιαία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ένα πολύ μεγάλο ειδικό βάρος και αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν αυτού όμως θέλω να πω ότι οι χώρες BRICS δεν έχουν τόσο μεγάλη σχέση μεταξύ τους, τόσο μεγάλη ομοιότητα είτε, ή τόσο μεγάλη συνεργασία μεταξύ τους όπως μπορεί να φαίνεται. Δρούν με τρόπο ο οποίος είναι πολλές φορές αποκλίνων και όχι ενιαίος. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να συνάψει εταιρικές σχέσεις με τις χώρες αυτές. Δεν βλέπω όμως την ανάγκη να υπάρξει μια ειδική στρατηγική για τις χώρες BRICS μέσα στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σας το λέω αυτό, γιατί κατά τη δική μου άποψη αυτές οι ομάδες δεν αποτελούν ένα μπλοκ παρά το γεγονός ότι έχουν ένα, μια ακροστοιχίδα, ένα όνομα που τις ενώνει όλες. Δεν αποτελούν ένα συνεκτικό σύνολο. Για όλους αυτούς τους λόγους θα έπρεπε να έχουμε συντονισμό της εξωτερικής μας πολιτικής μεν, αλλά δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σαν ένα ομογενές σύνολο της χώρας BRICS. να εστιαζόμαστε μόνο σε μία ή δύο χώρες μόνο, τις Ηνωμένε Πολιτείε ή κάποια άλλη χώρα. Σχετικά με την άποψη του δικού μας Κοινοβουλίου, πιστεύω ότι δεν χρειαζόμαστε να εκπαιδεύσουμε επιπλέον προσωπικό. Δεν χρειαζόμαστε πρόσθετο προσωπικό. Επίσης, έχω ένα ερωτηματικό σχετικά με τις προτάσεις αυτές, οι οποίες το μόνο που κάνουν είναι να αυξάνουν τη γραφειοκρατία και να την ενισχύουν. Ξέρετε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές εξωτερικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την εξωτερική πολιτική του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, του Συμβουλίου και έχετε εξωτερικές πολιτικές κατά τομέα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ομοιογενειοποίηση των εξωτερικών πολιτικών και ένα μόνο αριθμό του τηλεφώνου. Αρμόδιο. Η κυρία Γκόμες. Um, Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σάριος Βόλσκι για την έκθεση αυτή που καταδεικνύουν και το γεγονός ότι έχει λάβει υπόψη όλα τα σχόλια των συναδέλφων. Νομίζω ότι είναι πολύ θετική αυτή η αντιμετώπιση του και δείχνει ότι και η συζήτηση σε αυτή την Επιτροπή είναι χρήσιμη. Και εγώ Νομίζω ότι μπορώ να υποστηρίξω τα σχόλια του κυρίου Τσάλα, του σκιώδου συζητητή από τη δική μου πολιτική ομάδα. Απλώς θέλω να υπενθυμίσω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να μας κατευθύνει σε σχέση με την στάση μας για τις χώρες BRICS είναι να κατανοήσουμε ότι δεν είναι μια συνεκτική ομάδα. Μπορεί σε κάποιες στιγμές να υπάρχουν συνέργειες μεταξύ τους, αλλά αυτό το οποίο φέρνει τις χώρες αυτές από μαζί είναι μονάχα η ανάγκη μερικέ πληθών από εμά και να εναντιωθούν από σε εμά. Αλλά έχουν πολύ ουσιαστικέ διαφορέ μεταξύ του μέσα στην ομάδα αυτή. Εμεί τι ε, βάζουμε όλε τι χώρε αυτέ στο ίδιο καλάθι και αυτό είναι λαθασμένο. Υπάρχει πολλέ φορέ μια μεγάλη αντίφαση μεταξύ τους σε σχέση με τη στάση που κρατάνε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δύο από αυτές τις χώρες έχουν μια πολύ συντηρητική, μη μεταρρυθμιστική στάση, η Ρωσία και η Κίνα, θέλουν τη διατήρηση του status quo. Δύο άλλες, η Ινδία και η Βραζιλία, θέλουν να αποκτήσουν εκπροσώπηση ως μόνιμα μέλη στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτή είναι μία μείζον διαφορά, η οποία δεν πρέπει να παραγνωριστεί. και που θα πρέπει να αντανακλάται στις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόμαστε να ακολουθούμε πολλές φορές τη στάση της Ρωσίας και της Κίνας υπέρ του status quo Όλη η ρητορική λοιπόν για τη διεύνηση του Συμβουλίου της Ασφάλειας, της μεγαλύτερης νομιμοποίησης του Συμβουλίου Ασφαλείας, να, μην γίνεται, να γίνεται πιο αξιόπιστο το Συμβούλιο Ασφαλείας, όλα αυτά είναι αερολογίες. Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε δύο δυνάμεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μόνιμα μέλη, που δεν θέλουν καμία αλλαγή. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε εάν δεν υπάρχει αυτή η αύξηση αξιοπιστία του Συμβουλίου Ασφαλεία. Όλο και περισσότερο θα βρίσκεται σε αντίφαση το Συμβούλιο Ασφαλεία με την πραγματικότητα και αυτό υποσκάπτει τη δράση του. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο μα θα πρέπει να αναλάβουν το ρόλο του να ζητήσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια ενιαία θέση στο Συμβούλιο ασφαλεία, μια έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτό είναι αλλαγή του status quo και αυτό μπορούμε ίσως να το δούμε να αντανακλάται και στην έκθεση του κυρίου Σάριου Βόλφ και όταν μιλάει για τι χώρε BRICS. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Κρίστιαν Λεφλέ, ο οποίο είναι ε, διευθυντή ε, στην Υπηρεσία Εξωτερική Δράση με ιδιαίτερη αρμοδιότητα για την Αμερική. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να είμαι και εγώ εδώ για να σχολιάσω αυτό το σχέδιο της έκθεσης. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που το Κοινοβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις χώρες BRICS και στο ρόλο τους σε διεθνές επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια και κυρίως πέρυσι υπήρξαν πολλές συζητήσεις, ε, προβλήθηκε το θέμα των χωρών αυτών ε, στα μέσα ενημέρωσης, ε, προβλήθηκε το θέμα των χωρών BRICS και των αναδειωμένων δυνάμεων. Αυτή λοιπόν η ομάδα, στην οποία προστέθηκε πρόσφατα και το S της, ε, τα αρχικά της Νοτιοαφρικής, αυτοί από το 2009 συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πρέπει όμως ε, να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Ορισμένοι ε, βουλευτές επισήμαναν ήδη ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις χώρες αυτές ως ένα ομοιογενές μόρφωμα ε, μερικές φορές και το βλέπουμε αυτό και στις, ε, ε, στα ανακοινωθέντα τύπου μετά από συναντήσεις τους βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια διαφοροποίηση ως προς τους στόχους που επιδιώκουν. Νομίζω λοιπόν ότι οφείλουμε να αναλύσουμε προσεκτικά όλους τους τομείς, όλα τα θέματα το πώς ακριβώς συνεργάζονται, πού συνεργάζονται και ποιες είναι και οι διαφορές τους. Γιατί υπάρχουν ε, ε, κάποιες δράσεις ε, που τις ανέφεραν στα Ηνωμένα Έθνη, για άλλα θέματα συμφώνησαν, όχι όμως για όλα. Και δεν υπάρχει μόνο το στρατηγικό θέμα τη σύνθεση του Συμβουλίου ασφαλή. υπάρχουν και σημαντικά πολιτικά θέματα επί των οποίων δεν συμφώνησαν ή αν θέλετε ε, δεν κατέληξαν μέχρι τέλους στο να παραμείνουν συμφωμένοι. Παραδείγματο χάνει, για την περίπτωση τη Συρίας ε, συμφώνησαν για κάποιο χρονικό διάστημα μετά όμως ε, αντέδρασαν διαφορετικά το καθένα εξ αυτών όταν υπήρξε το καλοκαίρι μία αποστολή διαμεσολάβησης δεν είναι τυχαίο το ότι η Ινδία, Βραζιλία και Νότιος Αφρική, οι χώρες, μόνο αυτές οι χώρες αυτές πήγαν επιτόπου στη Συρία. Ενώ η Ρωσία και η Κίνα, για λόγους που έχουν άμεση σχέση με τα δικά τους συμφέροντα, δεν συμμετείχαν σε αυτή την αποστολή. Βεβαίως ε, θα μπορούσε κανείς ε, να αναφέρει ε, και τις, ε, τη στάση που κράτησαν στις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή και εκεί υπήρξε ουσιαστική διάσταση απόψεων μεταξύ τους. Ή, αν θέλετε, ε, τη δουλειά που γίνεται στην συνάντηση κορυφή στην G20 και εκεί υπάρχει διαφορά απόψεων. Νομίζω λοιπόν ότι ίσως θα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση για κάθε μία από τις χώρες αυτές. Έχουμε σημαντικές σχέσεις μαζί τους, θέλουμε να τις αναπτύξουμε περαιτέρω, επιθυμούμε να αναζητήσουμε τα κοινά στοιχεία και επιθυμούμε βεβαίως οποτεδήποτε λειτουργούν ως ομάδα να το δεχτούμε, να, να τους αντιμετωπίσουμε ως ομάδα. Όμως ε, δεν ε, είμαστε σε θέση, ούτε και μας συμφέρει και το να φροντίσουμε εμείς να τους ενώσουμε σε ομάδα. Έτσι λοιπόν, το να αντιμετωπίζει κανείς τις ε, χώρες αυτές ως νέες αναδυόμενες δυνάμεις αυτό θα σήμαινε όμως ότι αδικούμε μία σειρά άλλων πολύ σημαντικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν συμμετέχουν στην ομάδα αυτών των χαρών των BRICS που όμως ε, έχουν πολλές φορές ε, άμεσες σχέσεις με κάποιες από τις χώρες BRICS. Να αναφέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, την Τουρκία, το Μεξικό, την Κορέα, την Ινδονησία και πάρα πολλές άλλες. Και επιτρέψτε να φέρω και ένα σύντομο παράδειγμα. Όταν ο πρόεδρος Μαρούσεφ ε, ήρθε στις ε, Βρυξέλλες ε, πριν από ένα μήνα περίπου για τη συνάντηση κορυφής ή πρόεδρος, με συγχωρείτε, η πρόεδρος της Βραζιλίας ήρθε εδώ για την πρώτη συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επέλεξε τις Βρυξέλλες λόγω της σχέσης που υπάρχει με τη Βραζιλία, μετά Σοφία, Σόφια με και Βουλγαρία, γιατί έχει ρίσει από εκεί και κατόπιν πήγε στην Τουρκία. Γιατί για τη Βραζιλία η Τουρκία είναι ένα σημαντικό στρατηγικός εταίρος. Οφείλουμε λοιπόν να το έχουμε αυτό κατά νου οποτεδήποτε έχουμε σχέση με τη Βραζιλία αλλά και με την Τουρκία. Και οι πέντε χώρες της ομάδας BRICS είναι στρατηγικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δηλαδή τμήμα Ε, της πρωτοβουλίας ε, της κυρίας Άστον μετά από αίτημα του Συμβουλίου πριν από ένα περίπου χρόνο. Ο στόχος είναι να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα αυτή τη στρατηγική συνεργασία. Πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη σχέση με κάθε ένα εξ αυτών των εταίρων ε, και όπως σας είπα, οποτεδήποτε υπάρξει και ομαδοποίηση, πάρα πολύ ωραία. Εμείς λοιπόν πρέπει να αναζητήσουμε τους τομείς όπου υπάρχουν κοινά συμφέροντα, μπορούμε να δράσουμε από κοινού είτε σε πολυμερές επίπεδο είτε πιο συγκεκριμένα για συγκεκριμένα θέματα. Ήδη λοιπόν έχουμε πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδία για την αντιμετώπιση της πειρατείας στον Ινδικό ωκεανό. Έχουμε ε, ταχύτατα αναπτυσσόμενη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βραζιλία για αναπτυξιακά θέματα ε, εκτός Λατινικής Αμερικής, στην Νοτιοανατολική Ασία και στην Αφρική. Επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά παραδείγματα και ελπίζουμε στο μέλλον να υπάρξουν ακόμα περισσότερα για άλλες παρεμφερείς δράσεις. Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία συγκεκριμένα εσωτερικά θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση. Το ένα είναι στην παράγραφο υπαριθμών 5. Εκεί γίνεται λόγος για την ομάδα G20 ότι είναι το απόλυτο και κατάλληλο φόρουμ για να επιτευχθεί η συνένεση. Εμείς συμφωνούμε ότι η G20 είναι ένα πολύ σημαντικό φόρουμ, κυρίως για τους λόγους που αναφέρονται στην έκθεση. Ε, πρόκειται για μια νέα ομάδα κρατών ε, στην οποία συμμετέχουν ομάδες ε, χώρες BRICS αλλά και άλλοι σημαντικοί εταίροι που είναι εκτός ε, του παραδοσιακού κατεστημένου πλαισίου. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή την ομάδα, την G20, έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε κάποια θέματα ε, τα οποία κατά κανόνα ε, αν δεν λαμβάνουν χώρα εκεί αλλά σε παντοσιακό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα επίπονα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να αναζητήσουμε τη συνένεση με τις χώρες BRICS και άλλους εταίρους μας στην ομάδα των G20. Αλλά εγώ θα είμαι λιγάκι επιφυλακτικός. Δεν θα έλεγα ότι είναι το απόλυτο και μοναδικό φόρουμ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα φόρουμ όπως αυτά των Ηνωμένων Εθνών ή διεθνή χρηματοπιστωτικά φόρουμ και άλλα πλαίσια ε, πολύπλευρα και πολυμερή μέσα στα οποία επιθυμούμε να συνεργαστούμε με τις χώρες BRICS και με άλλες. Στην παράγραφο υπαριθμών 7 στην έκθεση υπογραμμίζεται η σημασία του συντονισμού της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την καθοδήγηση της ύπα εκπροσώπου. Αυτό λοιπόν ε, αφορά το άρθρο 21 και το άρθρο 26 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτά τα άρθρα προβλέπεται η απόδοση της απόλυτης αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ύπατη εκπρόσωπο για να μεριμνά αυτή για την συνέπεια των δράσεων της Ένωσης. Ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής η ύπατη εκπρόσωπος προσπαθεί να ε, βρει ε, την καλύτερη διασύνδεση της εξωτερικής πολιτικής με άλλους τομείς δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθεί να διασυνδέσει την εξωτερική πολιτική και με τομείς αρμοδιοτήτων άλλων συναδέλφων της στην Επιτροπή. Ως είπατη εκπρόσωπος και πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων προσπαθεί να επιφέρει μεγαλύτερη κινητοποίηση ε, σε διάφορες δραστηριότητες ε, που αφορούν στα κράτη-μέλη και αυτά αναζητώντας και επιδιώκοντας την επίτευξη κοινών στόχων που καθορίστηκαν από τους θεσμούς μετά από προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και που στηρίχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εμείς λοιπόν Χαιρετίζουμε την υποστήριξη αυτής της έκθεσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έννοια ότι διασφαλίζεται ο σημαντικός ε, συντονιστικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως ακριβώς προβλέπεται από ε, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ε, ΥΠΑ της Εκπροσώπου. Το τελευταίο που θέλω να πω κύριε Πρόεδρε αφορά στην παράγραφο υπαριθμών 9 στην έκθεση. Εκεί προτείνεται να συσταθεί μια ομάδα συντονισμού με την υπηρεσία, από εκείνο με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι χώρες BRICS ε, συστημικά θα είναι συμβατές. Εγώ λοιπόν θέλω να σας προειδοποιήσω, ε, να προειδοποιήσω να μην υπάρξει αυτή η ειδική μονάδα. Και ξέρετε γιατί, κυρίως διότι πολλοί από εσάς θα θυμάστε, αν ανατρέξουμε πίσω στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη σύσταση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο προβλήθηκε τόσο από το Συμβούλιο όσο και από το Κοινοβούλιο και συμφωνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα λοιπόν σημαντικό στοιχείο ήταν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο γεωγραφικό γραφείο. Που σημαίνει, αν έχουμε τώρα μια ειδική μονάδα για τις χώρες BRICS, αυτό μπορεί να προκαλέσει κάποια ένταση, ακόμα και σύγχυση. Σύγχυση για το ποιος τελικά φέρει την αρμοδιότητα. Ποιος είναι εκείνο που καθοδηγεί τις σχέσεις με την Κίνα, τη Βραζιλία, την Ινδία ή ακόμα και τη Νότια Αφρική. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι είναι καλύτερα την διαχείριση των σχέσεων με κάθε μία από τις χώρες αυτές να την αφήσουμε τη διαχείριση υπό την καθοδήγηση του εννέου γεωγραφικού γραφείου όπως αναφέρεται. Προβλέπεται αυτό στη σύσταση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και βεβαίως το γραφείο αυτό να στηρίζεται από τη μονάδα στρατηγικού σχεδιασμού που συστήθηκε και αυτή από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και έχει ως στόχο να ε, έχει το βλέμμα στραμμένο λίγο πιο βαθιά στο μέλλον από ότι το ε, πράττουν οι άλλες μονάδες που εργάζονται περισσότερο σε καθημερινή βάση. Αυτό που ενδιαφέρει επίση είναι μέσα στην ίδια την υπηρεσία εξωτερική δράση να υπάρχει ένα άτυπο δίκτυο, αν θέλετε, πέστε το Task Force, ομάδα κρούση. Αυτή η ομάδα μπορεί να συντονίζει τα διάφορα γραφεία που είναι αρμόδια για σχέσεις με τις χώρες BRICS ή με τους βασικούς στρατηγικούς εταίρους και από εκεί να προκύπτει ο απόλυτος συντονισμό, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τελικά πράγματι θα έχουμε μια συνεπή, συνεκτική προσέγγιση προς κάθε μία από τις χώρες αυτές. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρέμβασή σας. Και η τελική ε, κατακλείδα για να κλείσει η συζήτηση θα παρουσιαστεί από τον κύριο Σάιρου Βόλσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα βρίσκω ότι υπάρχει σύγκληση των απόψεών μου, των δικών μου και της κυρία Σάλα. Δεύτερο, για τα θέματα κλειδιά. Τα, τα γεγονότα είναι ως ε, εξής. Συναντώνται τακτικά, συντονίζονται, λαμβάνουν κοινέ δράσεις και μέτρα. Έχω έξι που ε, για την Λιβύη, για τα Ηνωμένα Έθνη, για την ακτή του Ελεφανταστού, για ε, το διάστημα, το Σουδάν και τη Συρία. Αυτά είναι γεγονότα και ακόμα και αν αυτά τα γεγονότα είναι 5% ε, του συνόλου ή ακόμα και 1% των BRICS δεν είναι λόγος για να μην αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν. Να διατηνόμεθα ότι δεν υπάρχουν. Και εδώ αναφέρομαι στην παρατήρηση του συναδέλφου από την ομάδα των Πρασίνων ότι θα έπρεπε ε, να τους θεωρήσουμε ως ανήλικες πρωταγωνιστές της παγκόσμιας κονίστρας, αντί να υιοθετούμε την άποψη ότι δεν έχουν μεγαλώσει, ότι δεν έχουν οριμάσει. Και λέγοντας αυτό, ε, θα έπρεπε να αποφύγουμε τέτοια συμπλέγματα απέναντι στους BRICS στην πολιτική μας και δεν έχουμε εμείς συμπλέγματα αυτού του είδους. Σχετικά με τις παρατηρήσεις ε, της, που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεν θεώρησα εγώ ότι, είναι η ομάδα αυτή είναι συνεκτική. Αντίθετα, ε, ορισμένες χώρες παρεκκλίνουν, υπάρχουν διχογνωμίες και τις οποίες ανέδειξα. Αναφερθήκατε στα τρία θέματα. Το πρώτο θέμα, παραγράφο 5 για τη G20, ναι, συμφωνώ πλήρω. είναι το φόρουμ όπου μπορούμε να συναντήσουμε τις χώρες αυτές. Για την παράγραφο 7 είπα ότι εκπρόσωπος, η δράση της ναι, βεβαίω, είναι στην συνθήκη, αλλά είναι αυτό μια πραγματικότητα. Έχει εφαρμοστεί αυτή η διάταξη της συνθήκης. Όχι, όχι επαρκώς θα έλεγα. Παραγραφό 9. Ε, ομάδα συντονισμού. Μιλάμε εδώ για μια ad hoc μονάδα συντονισμού. Οποιοδήποτε όνομα δώσουμε σε αυτήν την μονάδα, νομίζω ότι ήδη η έκθεση θα έχει παίξει καλό ρόλο ικανοποιητικό, διότι θα προετοιμάσουμε ε, την αντίδραση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης σε αυτήν την εισήγηση. Βεβαίως η Ινδία, η Κίνα δεν συναντώνται και δεν συνομιλούν μεταξύ τους. Είτε την ονομάσουμε αυτήν την μονάδα, ομάδα κρούσης, ομάδα δράσης ή ad hoc μονάδα συντονισμού, νομίζω όμως ότι είναι απαραίτητη, ανεξάρτητα από την ονομασία που θα της δώσουμε. Ε, ναι, καταλαβαίνω αυτήν την γεωγραφική προσέγγιση, αλλά μήπως αυτή είναι 19-20ου αιώνα ε, προσέγγιση. Ο κόσμος δεν είναι πια μια, ένα συνονθήλευμα υπήρων και μεγάλων μονάδων. Νομίζω λοιπόν ότι γενικά ήδη υπάρχει μια πρόοδος στη σκέψη μας και αυτό με ικανοποιεί ιδιαίτερα. Δεύτερον, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην μεταχείριση μεμονωμένων μη συνεκτικών ομάδων ε, και με συνεκτικό τρόπο σε ορισμένους τομείς. Μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις. Και αν κάποιος ε, είπε, νομίζω ότι ήταν η κυρία Γιατανμάκη, η οποία είπε ότι ότι είναι λιγότερο συνεκτική αυτή η ομάδα από ό,τι είμαστε εμείς. Ας πάρουμε το θέμα της Λιβύης. Ε, υιοθέτησαν μία ενιαία θέση απέναντι ε, στην Λιβύη χωρίς δομές, χωρίς μονάδες ιδιαίτερες. Στην περίπτωση λοιπόν της Λιβύης, αυτή η ομάδα, η μη συνεκτική των BRICS, είχε αντιμετώπιση πιο συνεκτική από ό,τι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην υποτιμούμε λοιπόν το φαινόμενο των BRICS, ναι, τα όσα είπε η Άννα Γκόμες. Η τελική μου το τελικό μου συμπέρασμα είναι ότι χρειαζόμαστε μια έκθεση, μια ξεχωριστή έκθεση σχετικά με τις στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις. Δεν συμφωνώ με την προσέγγιση που εφαρμόζεται, υιοθετείται από την Ένωση και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ότι ό,τι είναι σημαντικό πρέπει ε, να ε, έχει στρατηγική. Ας δούμε τι είναι σημαντικό, υπερσημαντικό, αλλά ε, πρέπει να δούμε για την συνεργασία, τη μέση συνεργασία, να δούμε ποιε είναι οι δικέ μα οι αξίε. Η Βραζιλία είναι στρατηγική χώρα, διότι είναι δημοκρατία. Η Ινδία είναι στρατηγική χώρα. Η Ρωσία και η Κίνα είναι στρατηγικέ χώρε, ε, διότι ε, αυξάνουν τι ανησυχίε μα, τι στρατηγικέ και τι ελπίδε μα, αλλά δεν είναι στρατηγικέ διότι δεν συνεργάζονται καλά μαζί μα, διότι έρχονται σε αντιπαράθεση μαζί μα. Αμφισβητούν τη γλώσσα μα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κλιματική αλλαγή και ό,τι αφορά την δημοκρατία. Και απευθύνομαι στον πρόεδρο. Χρειαζόμαστε μια έκθεση για τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις και δεν πρέπει να αποφεύγουμε να αναγνωρίζουμε νέα γεγονότα στη διεθνή κονίστρα. Διότι είχαμε γεωγραφική εξωτερική πολιτική και εξακολουθούμε να έχουμε αυτήν την πολιτική ενώ ισχυριζόμεστα ότι ε, δεν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Αυτή είναι ψευδοπροσέγγιση. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια καλύτερη κατανόηση και μια συνένεση στην Επιτροπή μας σχετικά με αυτό, χάρη σε αυτή τη συζήτηση ε, και νομίζω ότι θα πρέπει και εμείς να δούμε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ποια είναι η προσέγγιση. Ίσως δεν ξέρω ένας καφέ στο διάδρομο με αυτούς τους ανθρώπους ξεχωριστά, τη Ρωσία, την Κίνα, την Βραζιλία, να τους συναντούμε, συναντούμε μια φορά το μήνα και να σκεφτούμε ε, ανεξάρτητα από το αν είναι στρατηγική ή μη στρατηγική εταίροι, να δούμε τι σκέφτονται και πώς, ε, ποια είναι η στάση τους απέναντι μας. Διότι την ώρα υπάρχει ένα χάσμα και ακόμα και αυτό το χάσμα είναι 1% της ε, ομάδας, της, της εικόνας 100%, ακόμα και αυτό το 1% έχει τεράστια σημασία, διότι έχουν, επηρεάζουν την ύπαρξή μας, την δυνατότητα να μιλούμε με μία φωνή. Βλέπουμε τη θέση που έλαβαν σε σε σχέση με τη Λιβύη. Ας ε, ξεχάσουμε μια μεγάλη δύναμη που ήταν στο περιθώριο, αλλά στο μέλλον. Εγώ ε, προβλέπω ότι το φαινόμενο αυτό θα ενισχυθεί και δεν θα μειωθεί. Συνεπώς, η πολιτική του να μην αναγνωρίζουμε την ομάδα, αυτή την πολιτική του στρούθοκαμιλισμού, δεν είναι καλή γραμμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα όσα είπατε για την ποικιλομορφία, για τις αντιτεθέμενες απόψεις και συμφέροντα, την ανάγκη να ασχοληθούμε ξεχωριστά με μονεμένα με κάθε χώρο, όλα αυτά είναι σωστά, αλλά μην ξεχνούμε αυτόν τον συντονισμό που αυξάνεται, που ενισχύεται μεταξύ των χωρών της ομάδας, δεν ξέρω πώς θα τον ονομάσουμε ονομάσουμε και θα πρέπει από δική μας πλευρά να έχουμε μια μέθοδο ανοιχτού συντονισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Α, μισό λεπτό. Να σας υπενθυμίσω ότι η ψηφορία θα λάβει χώρα στις 20 Δεκεμβρίου. Επόμενο θέμα είναι η έκθεση του κυρίου Παντσέρη, Προέδρου της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέπ σχετικά με την 11η Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Αλγερίας, μια συνάντηση που έλαβε χώρα από τις 2 μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στο συνάδελφο ε, κύριο Παντσέρη για να μας ε, παρουσιάσει τα θέματα που συζητήθηκαν με τις αρμόδιες αρχές και θα ήθελα κυρίως ε, το δικό του σχόλιο για τρία θέματα. Το πρώτο είναι η τρέχουσα κατάσταση, η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Αλγερία από το πρίσμα της εθνικής και της περιφερειακής ασφάλειας. Δεύτερον, την άποψη των αρχών της Αλγερίας για αυτά που διαδραματίζονται στις χώρες Μαγκρέμπ και Τρίτον, τρίτο σημείο, τις ε, αντιδράσεις ε, που διαπιστώσατε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας για το ενδεχόμενο να υπάρξει στο μέλλον Επιτροπή Παρακολούθησης Εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλγερία. Ο κύριος Παντσέρη έχει το λόγο. Όπως είπατε, η συνάντηση έλαβε χώρα από τις 2 μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Η δική μας λοιπόν η αποστολή είχε ως ε, γενικούς στόχους ε, να εξετάσει, να αξιολογήσει τη βούληση πολιτικών μεταρρυθμίσεων μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ε, Αραβικής Άνοιξης, κυρίως όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες και στις εκλογικές διαδικασίες. Επίσης, να αξιολογήσουμε το νόμο περί ε, συνελεύσεων, περί, το νόμο του συνέρχεστε. Κατόπιν, θα θυμάστε ότι υπήρξε μια επιτροπή ε, παρακολούθησης ε, προτείναμε να υπάρξει Επιτροπή Παρακολούθηση Εκλογών όπως έγινε και στην Τινησία. Και είχαμε και άλλο ένα στόχο, ο οποίος ήταν να προτείνουμε τη θέσμηση ενός ειδικού οργάνου δύο αρμόδιων αρχών σε επίπεδο Αλγερίας. Η μία να αφορά τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και τέλος να ενθαρρύνουμε τις αρχές της Αλγερίας να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την εφαρμογή ενός προγράμματος δράσης. Εδώ λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ε, συναντήθηκε με ορισμένους ε, θεσμικούς ε, εκπροσώπους, με τους δύο εκπροσώπους της Άνω και Κάτω Βουλής, με τον Πρωθυπουργό, Υπουργό Εξωτερικών, τον εντεταλμένο Υπουργό για τις σχέσεις με τις χώρες Μαγκρέπ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας είχαμε μία συζήτηση με το Κοινοβούλιο που αποτελείται από τους βουλευτές ε, που εκπροσωπούν τις διάφορες περιοχές. Ε, στο πλαίσιο των συζητήσεων ετέθη το θέμα τη συνεργασία. Αυτό με ενδιαφέρει και τι δύο πλευρέ, δηλαδή η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτικέ μεταρρυθμίσει που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή, η κατάσταση στην Αλγερία κάτω από το πρίσμα το, του ευρύτερου χώρου του Μαγκρέμπ. Οι βουλευτές Αλγερίας παρουσίασαν στη δική μας την Επιτροπή την διαδικασία πολιτικών μεταρρυθμίσεων που λαμβάνει η χώρα στην Αλγερία και επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ε, ολοκληρώσουν αυτό το δρόμο. Είπαν επίσης ότι θέλουν να εμβαθύνουν στις δημοκρατικές διαδικασίες, να υπάρχουν περισσότερες πολιτικές ελευθερίες και να προβλέπεται καλύτερη διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή επίσης ενημερώθηκε για την οικονομική συγκυρία στην Αλγερία και για τις προοπτικές που υπάρχουν στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των συζητήσεων, οι δύο αντιπροσωπείες κατέληξαν στα εξή ε, κοινά συμπεράσματα και αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν δύσκολο να βρούμε σημείο επαφής με, τους, ε, με το Κοινοβούλιο της Αλγερίας. Πρώτον, εκείνο που υπογραμμίσαμε και οι δύο πλευρές ε, είναι ότι υπάρχει εξέλιξη των σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αλγερία μετά την θέση σε ισχύ ε, της ε, Συμφωνίας σύνδεση. Το 2005 έγινε αυτό. Υπάρχει λοιπόν στρατηγικός χαρακτήρας του διακοινοβουλευτικού διαλόγου και είναι απαραίτητο αυτό να ενισχυθεί περαιτέρω, να υπάρχει πιο στενή συνεργασία Αλγερίας ε, και Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της νέας πολιτικής γειτονίας. Επίσης υπογραμμίστηκε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μία μόνιμη επιτροπή με το ε, Κοινοβούλιο της ε, Αλγερίας και με τις δύο βουλές. Αυτό θα συμβάλλει στην βελτίωση των σχέσεων Μαγκρέμπ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έτσι θα συνεχιστεί και ο πολιτικός διάλογος. Οι πολιτικέ μεταρρυθμίσεις αποτελούν μία μοναδική ευκαιρία και αυτό αυτό αφορά την έγκριση του νόμου για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή. Ε, αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο και πρέπει να προχωρήσει από κοινού με την συμμετοχή των γυναικών ε, στην οικονομική και κοινωνική ζωή, κυρίως με δράσεις που να αφορούν στην πρόσβαση στην απασχόληση. Πρέπει λοιπόν ε, να υπάρξουν ε, συνομιλητές από πλευράς Αλγερίας, ε, κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο. Η ελευθερία του συνέρχεται πρέπει να είναι απόλυτα διασφαλισμένη δική μας η ε, χρηματοδότηση θα γίνεται με τρόπο διαφανή. Όσον αφορά την κατάσταση περιφέρειας υπογραμμίστηκε ότι οι χώρες ε, Μαγκρέμπ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία, κυρίως όσον αφορά την Ένωση Μεσογείου. Η περιφερειακή συνεργασία πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω με απότερο στόχο τελικά να εξευρεθεί μια ικανοποιητική λύση στις περιφερειακές προκλήσεις. Η αποφασιστικότητα των αρχών Αλγερίας για να διασφαλίσουν ότι οι νομοθετικές διατάξεις που θα λάβουν χώρα για το 2012, ότι οι διατάξεις αυτές και οι διαδικασίες θα είναι διαφανείς και ελεύθερες, αυτό το εκτιμήσαμε ιδιαίτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε την μεγάλη της εμπειρία στην Αλγερία, ε, κυρίως όσον αφορά την παρακολούθηση εκλογών και δήλωσε ότι ε, αν θέλει η Αλγερία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την εμπειρία, κυρίως ε, ας μην ξεχνάμε ότι υπήρξε και αυτή η συζήτηση ήδη σε, παλαιότερα σε διάρκεια αυτού του έτους. Ο πρόεδρος Αλμπερτίνη και Ζολή ε, μπορούν να ε, παρακολουθήσουν τις εκλογές έτσι ώστε για να αποφευθούν καταστάσεις ανασφάλειας που θα μπορούσαν να θέσουν σε ε, κίνδυνο την όλη διαδικασία. Εμείς λοιπόν επιμένουμε ότι ε, όταν κάνουμε παρακολούθηση εκλογών είτε γίνεται όπως έγινε στην Τινησία είτε αλλιώς είναι καθαρά για τουρισμό. Τέλος, τα μέλη ενθαρρύνουν ε, να καταργηθούν οι δασμοί, να εξευρεθεί μια λύση στο πλαίσιο της ε, συμφωνία που υπάρχει και αυτή η συμφωνία είναι εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν. Προφανώ λοιπόν έχουμε και την ε, συμφωνία που αφορά στην κοινωνία των πολιτών. Αυτέ οι συναντήσει ήταν ιδιαίτερα σημαντικέ γιατί κατέστησαν ε, σαφέ ε, το ποιε είναι οι σχέσει που υπάρχουν με την Αλγερία και τι δυσκολίε που υπάρχουν σε επίπεδο κοινωνία των πολιτών. Τέλο, θα μου επιτρέψετε να καταθέσω κάποιε προτάσει να δώσω και κάποιε πληροφορίε ήδη ε, ε, με, με επιστολή ενημερώσαμε τον πρόεδρο κύριο Αλμπερτίνη αλλά θέλω και εδώ να επαναλάβω ορισμένα σημεία. Σας ενημερώσαμε για την επιστολή που αποστήλαμε στον πρόεδρο της Υποεπιτροπής ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με μια συνεδρίαση που να αφορά ε, στα δικαιώματα των ε, προσφύγων από τις χώρες Μαγκρέμπ. Όσον αφορά τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει μια κοινή συνεδρίαση της ΑΦΕΤ άλλων φορέων και των χωρών Μαγκρέμπ για να αντιμετωπιστεί το σημαντικότατο θέμα που είναι η περιφερειακή συνεργασία μεταξύ Αλγερίας, και άλλων χωρών ε, για να ε, συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το διάλογο, σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό το συζήτησε και η δική μας αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια της ε, συζήτησης, συνάντησής μας με τον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών της Αλβερίας που έχει επίσης υπό την αρμοδιότητά του και τις σχέσεις με τις χώρες Μαγκρέπ. Αυτή την επιστολή θα την στείλουμε και στις δύο βουλές της Αλγερίας έτσι όπως σας είπα να υπάρξει τελικά ένα θεσμικό όργανο το οποίο να επιλαμβάνετε των σχέσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας πω, η Επιτροπή, αυτή η αποστολή Μαγκρέπ της οποίας και προείσταμε, θα έχει επαφές με τους ε, επιχειρηματίες, αυτό είναι το ανεπίπεδο και το άλλο επίπεδο με τις οργανώσεις νέων. Και να πω ότι με την ευκαιρία της επαιτίου της ε, ανεξαρτησίας της Αλγερίας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να οργανωθεί μια φωτογραφική έκθεση ε, και τέλος επιτρέψω να φέρω και άρα δύο σημεία τα οποία θεωρώ σημαντικά. Όσον αφορά την Δυτική Σαχάρα είχα την ευκαιρία, επειδή ήμουνα στην Αλγερία, είχα λοιπόν την ευκαιρία να επισκεφθώ το Κιντούφ και ε, με συγχωρείτε. Και θεωρώ ότι πρέπει να ε, προβάλλουμε και πάλι τις σχέσεις ε, που προβλέπονται από τις τρεις μας επιτροπές και επίσης προτείνω στις 28 και 29 Νοεμβρίου να μεταβούμε στα Ηνωμένα Έθνη. Η τα ανθρώπινα ανθρωπιστικέ συνθήκες είναι ανησυχητικέ, όπως ε, και η χρήση με την οποία, η χρήση της ε, βοήθειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να εξεταστούν από την Επιτροπή μας. Είναι λοιπόν σημαντικό όσον αφορά του ε, Πολυσάριο ή Πολυσάριο να προσκληθούν σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων με τις χώρες Μαγκρέπ. Και τέλος είχαμε και ένα προφορικό αίτημα ε, το οποίο σας το μεταφέρω όπως μου αναφέρθηκε από τους Σαράουι έτσι ώστε να ε, λάβει επιτόπου επίσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αξιολογηθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στους καταβλισμούς. Αυτά όσον αφορά την αποστολή την οποία οργανώσαμε στην Αλγερία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, ευχαριστούμε κύριε Παντσέρη. Πρόεδρε Παντσέρη, συγγνώμη. Κάποιος θέλει να λάβει το λόγο. Η κυρία Μπέναραμπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ήμουν μέλος της αποστολής στην Αλγερία για να απαντήσω στις ερωτήσεις που θέσατε κύριε Πρόεδρε σχετικά με τη σημερινή κατάσταση. Πρόκειται για μια κατάσταση όπου υπάρχει ισχυρή βούληση μεταρρύθμισης πολιτικής. Υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι που ψηφίζονται Σχετικά με το ποσοστό των γυναικών, την ποσόστοση των γυναικών, είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένας νόμος που ψηφίστηκε ούτως ώστε σε 20% των καταλόγων ε, οι γυναίκες να καλύπτουν 20% των καταλογών στις μικρές πόλεις, 30% στις μεσαίες πόλεις και 40% στις μεγάλες πόλεις, Αλγέρι, Οράν κλπ. και 50% για τους Αλγερινούς στο εξωτερικό. Αλλά νομίζω ότι οι ποσοστώσεις δεν αρκούν διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα που τονίστηκε από πολλές ε, ΜΚΟ και φεμινιστρίες. Υπάρχει το πρόβλημα της οικογένειας που υποχρεώνει ε, τις γυναίκες να ζητήσουν την άδεια για να κυκλοφορούν. Η ποσόστοση βεβαίως είναι μια πρόοδος, αλλά το θέμα του οικογενειακού κώδικα στην Αλγερία είναι σημαντικό, ούτως ώστε οι γυναίκες να μπορούν να δρουν τελείως ελεύθερα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονιστεί αυτό. Έθεσα την ερώτηση στον ε, πρόεδρο του Κοινοβουλίου που μου είπε ότι για την ώρα το οικογενειακό κώδικα δεν βρισκόταν στην ατζέντα των συζητήσεων σχετικά με την ασφάλεια. Για να τελειώσω, ένα άλλο θέμα που μου φαίνεται σημαντικό, ο κύριος Παντζέρη το ανέφερε, υπάρχει ε, ένα θέμα αρκετά σημαντικό είναι ένα σχέδιο νόμου που ακόμα δεν ψηφίστηκε. Νομίζω ότι ε, έχει ε, θα καθυστερήσει η ημερομηνία της ψήφισης σχετικά με τις οργανώσεις της ο πρόεδρος, κ. Μουσασί, του Συνδέσμου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έλαβε θέση ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διότι το νόμο σχέδιο μπορεί να πνίξει κατά κάποιο τρόπο τις ε, οργανώσεις. δεν υπάρχει ένα πρόβλημα χρηματοδότησης. Θα χρειάζεται αδειοδότηση προτού δημιουργήσει κανείς μια οργάνωση. Πάρα πολλά σημεία αυτού ε, του νομοσχεδίου για τις οργανώσεις ε, κινδυνεύουν να πνίξουν τις οργανώσεις αυτές και οι ΜΚΟ είναι αρκετά ανήσυχες και ο κύριος Μουσασί, πρόεδρος του Συνδέσμου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είπε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε σχέση με το νομοσχέδιο αυτό. Δεδομένου ότι η ημερομηνία αυτή έχει αναβληθεί, ελπίζουμε να υπάρξει πρόοδος σε σχέση με το θέμα αυτό. Σε σχέση με την ασφάλεια στο Μαγκρέμπ και στην Αφρική, ο Υπουργός ε, Αφρικανικών Υποθέσεων και Υποθέσεων του Μαγκρέμπ ε, μας μίλησε και ήταν σημαντική αυτή η συνάντηση διότι ο Υπουργός Μπεσαλέρ έχει μια θεώρηση, μια πραγματική στρατηγική σχετικά με την ασφάλεια. Υπάρχει μια ομάδα που δημιουργήθηκε με, τα, με τις πέντε χώρες του Σαχέλ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Βρίσκω ενδιαφέρον να ε, υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική που ασχολείται ταυτόχρονα με ασφάλεια, άμυνα και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και καταπολέμηση της φτώχειας. Νομίζω ότι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ενώ θα υπάρχει πτώχεια, ο κίνδυνος ε, υπάρχει οι πολίτες ε, να να υιοθετήσουν θέσεις ακραίες για δράσεις που χρηματοδοτούνται σχετικά με την Επιτροπή Παρακολούθησης των Εκλογών. Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση για το θέμα αυτό. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε επανειλημμένα αν θα μπορέσουμε να έχουμε ε, μία αποστολή παρακολούθησης ε, των εκλογών εκεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναβλήθηκε η συζήτηση και τελικά μας είπαν ότι ε, θα υπάρξει μια πρόσκληση, ότι υπήρξαν όμως αντιθέσεις και υπήρξαν πρόεδροι κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του Αρσεντέ, ο Γενικός Γραμματέας, δεν ξέρω ποιος είναι ο τίτλος του, και εγώ συνήντησα τον πρώτο γραμματέα του FFS, δηλαδή του κόμματος της αντιπολίτευσης, που μου είπαν ότι ήταν αρκετά ανήσυχοι και ότι αυτή η βούληση, η δεδηλωμένη βούληση προς έναν εκδημοκρατισμό δεν τους πείθει και ότι υπάρχει ένας κίνδυνος η δική μας η Επιτροπή να χρησιμοποιηθεί από ΜΚΟ και ίσως να, δώσει, να αποτελέσει κάποια ίγκριση σε μια διαδικασία που δεν οδεύει πραγματικά προς τον εκδημοκρατισμό. Κάναμε σύγκριση με τα όσα συνέβησαν στην Τινησία. Η διαφορά με την Τινησία, και αυτό είναι σημαντικό να λεχθεί, είναι ότι υπήρξε μια επιτροπή ανεξάρτητη που οργάνωσε αυτήν την εκλογική διαδικασία και είχαμε τον υπεύθυνο ο οποίο ήταν αναγνωρισμένο, ενώ στην Αλγερία δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιτροπή. Θα είναι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνη, του Υπουργείου Εσωτερικών που θα οργανώσουν τι εκλογέ. και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα, η ανεξαρτησία αυτών που θα οργανώσουν τι εκλογέ. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα ε, ταυτόχρονα μας προειδοποίησαν, πρέπει βεβαίως να συμμετέχουμε, αλλά μας προειδοποίησαν ότι ως Ευρωπαίοι δεν πρέπει να εγκρίνουμε μια διαδικασία που μπορεί να αμφισβητηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να διευκνήσω δύο πράγματα. Όσον αφορά την στρατηγική ασφάλειας, εμείς ζητήσαμε κατηγορηματικά από την Αλγερία να προσπαθήσει να συμπεριλάβει και το Μαρόκο στον αγώνα κατά της ε, τρομοκρατίας, γιατί αυτό είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα και λεπτά θέματα. Ε, και αυτό πρέπει να γίνει, γιατί αυτό το οποίο διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή είναι πράγματι ιδιαίτερα περίπλοκο. Δηλαδή, απαγωγές που γίνονται στους καταπλησμούς Σαράουι, το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήγουν πουθενά από το πρίσμα της ε, Δυτικής ε, Σαχάρας, αυτά όλα θα οδηγήσουν κατά πάσα πιθανότητα σε ακόμα πιο ε, ριζοσπαστικοποίηση των δράσεων. Το γεγονός λοιπόν ότι εμείς, μάλλον το ότι υπάρχει και ουσιαστική παρουσία της Αλκάιντα σε αυτή την περιοχή και το γεγονός ότι υπάρχουν και όπλα που έρχονται από τη Λιβύη, όλα αυτά οδηγούν στο ότι πρέπει να συμμετέχουν και οι δύο χώρες στις συζητήσεις ε, με την τετραμερή. Να συμμετέχει οπωσδήποτε και το Μαρόκο. Τέλος, όσον αφορά την παρακολούθηση εκλογών. Το λέω ακόμα και αν δεν αρέσει σε κάποιους. Κοιτάξτε, ε, υπάρχουν πάρα πολλές χώρες ε, που πάνε για παρακολούθηση εκλογών σε αυτές τις περιοχές για δικά του συμφέροντα και δεν έχει καταλάβει κανείς εκπροσωπούν και δημιουργούν προβλήματα. Μερικοί λένε ότι, είναι, ότι παρακολουθούν τις εκλογές, άλλοι λένε ότι είναι φίλοι της χώρας. Κατά κάποιον τρόπο θα ήταν χρήσιμο πριν καταλήξουμε να υπάρχει μια πειθαρχία σε αυτές τις ε, επισκέψεις. Σας είπα, αν υπάρξει παρακολούθηση εκλογών να είναι πανομοιότυπη όπως έγινε και στην περίπτωση της Τινησίας. Και Επίσης ε, είχα μια συζήτηση με τον Επίτροπο κ. Φούλε και του είπα η Επιτροπή να έχει αυτή ακριβώς την διαστάση. Γιατί αν θέλουμε να πηγαίνουμε σε παρακολούθηση εκλογών πρέπει να είμαστε σοβαροί. Να αποφύγουμε ε, την ε, κατάτμιση της κοινωνία των πολιτών, να μην δημιουργήσουμε προβλήματα, αλλιώς να μην πηγαίνουμε καθόλου εκεί. Γιατί δεν νομίζω ότι αν δεν υπάρχουν αυτές οι εγγύησεις νομιμοποιείται οποιοδήποτε να πηγαίνει σε αυτές τις αποστολές. Ε, θα μου επιτρέψετε και εγώ να προσθέσω μια ερώτηση προς εσάς πρόεδρε Παντσέρη. Γνωρίζουμε πολύ καλά τη διαμάχη ανάμεσα στην Αλγερία και το Μαρόκο σχετικά με την, ε, την περιοχή Σαράουι. Αυτή τη στιγμή ποια είναι, ποιες είναι οι σχέσεις ανάμεσα στην Αλγερία και το Μαρόκο. Είναι καλές οι σχέσεις είναι ικανοποιητικές, ε, τέλειες, καταπληκτικές, ε, χάλια. Ε, ποιες είναι οι προοπτικές για το εγγύς μέλλον, τουλάχιστον όσον αφορά ορισμένα θέματα, παραδείγματος χάνει την τρομοκρατία και τον έλεγχο των συνόρων. Κύριος Παντσέρη, Κοιτάξτε, πέρα από αυτά που λένε στι επίσημε συναντήσει, οι σχέσει δεν τι χαρακτήριζα εξαιρετικέ. Υπάρχει πρόβλημα τόσο όσον αφορά τα οικονομικά και κοινωνικά θέματα όσο και τον αγώνα κατά της ε, τρομοκρατίας. Νομίζω η Αλγερία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να έχει τη δική της την υγειοπολιτική στάση, κυρίως στην περιοχή Σεχέλ και προσπαθεί κατά κάποιον τρόπο να αποκλείσει το Μαρόκο. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να διασφαλίσουμε τη συνεργασία γιατί με τον τρόπο αυτό θα έχουμε και τη συμμετοχή του Μαρόκου. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στις 11 ε, και 4, σε 20 περίπου λεπτά, θα έχουμε συνεδρίες και κλεισμένων των θυρών και θα έχουμε και ανταλλαγή απόψεων με τον ε, κύριο Ιωάο Κραβίνιο, ο οποίος είναι προσφάτως οριστής σε επικεφαλής αντιπροσωπής Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ινδία. Θα κάνουμε διάλειμμα για 20 λεπτά και θα επανέλθουμε στις 11 και 4 και κλεισμένο των θυρών. Σας ευχαριστώ.